σε μια κοινοβουλευτική, ε, για αντιπροσωπεία. Θα δημοσιευθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης. Αν μέχρι την έγκριση των πρακτικών δεν υπάρξει ένσταση, τότε θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται.